και η συνεδρίαση της Ολομέλειας, αφού σας πω όμως ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι αύριο 17 Ιουλίου από τις 10 μέχρι τη 1. Η ημέρησια διάταξη έχει διατυπωθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη συνεδρία και καλό βράδυ σε όλους και όλες.